Mes chers collègues, la séance est ouverte. Le groupe social... Αγαπητοί συνάδελφοι, αρχίζει η συνεδρίαση. Οι σοσιαλιστές κατέφθασαν και έτσι είμαστε έτοιμοι να ψηφίσουμε. Hopefully, hopefully. Hopefully. Je voudrais, euh, pendant que... Euh... Θα ήθελα, ενώ ετοιμάζεται η συγγήτρια, και φτάνουν και τελευταίοι καθυστερημένοι και ενώ όλοι παληθεύουν ότι έχουν ε, την κάρτα ψηφοφορίας τους, την ηλεκτρονική κάρτα και όλοι επαληθεύουν πως έχουν ε, όλους τους ψηφοφόρους τους, αλλά όχι υπερβολικά πολλούς. Να χαιρετήσω την παρουσία του κυρίου, της κυρίας Αντερζονάς, ζητώ συγγνώμη για την προφορά μου, που είναι πρόεδρος της Επιτροπής ε, Προϋπολογισμού και Οικονομίας του Κοινοβουλίου του Κωσυφοπεδίου και που είναι σήμερα εδώ. Και έχοντας μάθει από τον Ράιμερ Μπέγκη πως έχουμε αυτή τη συνεδρίαση, θέλησε να έρθει να παρακολουθήσει Εξ ονόματος της Επιτροπής Προπολογισμών, λοιπόν, κυρία Πρόεδρε, αγαπητοί συνάδελφοι, σας χαιρετίζω, σα ε, καλωσορίζω, Μα τιμά η επίσκεψή σας. Euh, Και καλή τύχη στο Κωσυφοπαίδιο. Chers amis, chers amis, alors, conformément à ce que nous avons... Αγαπητοί φίλοι, σύμφωνα με τα όσα αποφασίσαμε σήμερα το πρωί, τις ψηφοφορίες, ο κύριος ε, Γκάιρ Και θα ξεκινήσουμε από την κατηγορία 1β. Έχετε όλοι το κατάλογο ψηφοφορία σας. Comme Tout le monde a son, tout le monde a son tableau de vote. Est-ce qu'on peut commencer maintenant? Έχετε όλους τους καταλόγους ψηφοφορίας. Ωραία, ας ξεκινήσουμε. Κατηγορία 1β. Στο φύλλο μου είναι η σελίδα 88 του πίνακα. Το έχουμε όλοι στα αγγλικά. Είμαστε στην 88. Αρχίζουμε με την τροπολογία 41-25 του κύριου Χαρτόγκο. Η συγκεκριτής είναι κατά, ποιοι υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Στην επόμενη γραμμή έχουμε μια σειρά τροπολογιών που είναι ταυτόσιμες. Οπότε ψηφίζουμε την τροπολογία 405. Ο εισηγητής είναι υπέρ. Ποιοι είναι υπέρ. Κατά. Ευχαριστώ. Αποχές. Ε, το 405 ή 405 και οι υπόλοιπε 4 που είναι ταυτόσιμες εγκρίνονται. Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο. Τροπολογία 1 Αρτόγκ. Είναι η 4126 του κ. Αρτόγκ η συγκίτρια είναι κατά, υπέρ, αποχές απορρίπτεται. Η δεύτερη έχει αποσυρθεί. Η τροπολογία 751 είναι μια επιφύλαξη, είναι αποθεματικό, θα το ψηφίσουμε μετά. Το 10-11 θα ψηφίσουμε, η συγκίτρια είναι κατά, ποιον υπέρ. Κατά, αποχές, απορρίπτεται. 423. Η την υπέρ. Κατά. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Οι σοσιαλιστές βρίσκονται μόνοι τους. 714. Ποιοι είναι υπέρ. Κατά. Αποχές. Ίδια πλειοψηφία. Απορρίπτεται. Επανέρχομαι λίγο πιο πάνω, στην 751, γιατί πρέπει αυτό να μπει σε αποθεματικό. Είναι από τους πράσινους, η συγγήτρια είναι κατά. Ποιοι είναι υπέρ. Η πράσινη. Η... Ποιοι είναι κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 47-55 ψηφίζουμε τώρα για τις παρατηρήσεις. Η συγκίτρια είναι υπέρ. Ποια είναι υπέρ. Κατά. Αποχές, οι παρατηρήσεις συγκρίνονται. Στην 47-77. Υπάρχει ένα σχόλιο, αλλά με προφορική τροπολογία του κυρίου Σουριάν που σας έχει δοθεί. λέει ότι αυτά τα κονδύλια στηρίζουν βελτιώσει στην φροντίδα των παιδιών ώστε να διευκολυθούν τα παιδιά να ζουν στο οικογενειακό περιβάλλον. Σε οικογενειακό περιβάλλον. Το υπόλοιπο μένει το ίδιο. Ποιοι είναι υπέρ. Κατά. Αποχές. Νομίζω ότι απορρίπτεται. Αλλά θα το επαληθεύσουμε. θα ελέγξουμε ηλεκτρονικά. Εγώ μπορώ να ψηφίσω. Ψηφίζουμε. Ψηφίστε, ψηφίστε. Τέλος ψηφοφορίας. Ένας δεν έχει ψηφίσει. 18, 18. Απορρίπτεται. Ωραία. Γυρνάμε σελίδα. Δύο πρώτες τροπολογίες, 45-19, έχουν αποσυρθεί. Και ψηφίζουμε στη 41-27 του κυρίου Αρτόγκ, η συγγύτρια είναι κατά, ποιοι είναι υπέρ. Κατά. Αποχές, απορρίπτεται. Το επόμενο είναι ένα αποθηματικό, θα το ψηφίσουμε αργότερα. 424 τώρα, ποιοι είναι υπέρ, η συγγύτρια είναι κατά. Ποιοι είναι κατά. Αποχές απορρίπτεται. Οι δύο επόμενες τροπολογίες, η 934 και η 4687, όσον αφορά τις παρατηρήσεις, είναι μια αιτιολογία και όχι σχόλιο. Οπότε κατά τη γνώμη μου δεν χρειάζεται να ψηφίσουμε. Πρέπει να ψηφίσουμε για τα νούμερα. Να έχει νούμερα. Όμως ψηφίζουμε τις τροπολογίες που πάνε μέχρι το τέλος της σελίδας και στην 4307 του Κλάουντιο Μοργάντη που αντιστοιχούν στους ίδιους αριθμούς η συγκήτρια είναι υπέρ. Ποιοι είναι υπέρ αυτών των τροπολογιών κατά αποχές, δεν υπάρχουν αποχές. Μέχρι το τέλος λοιπόν εγκρίνεται. εγκρίνονται. Περνάμε στην επόμενη σελίδα, σε 41-28 αρτόγκ. Η συγκεκριμένη κατά ποιοι υπέρ. Α, με συγχωρείτε, με συγχωρείτε. Είμαι υποχρεωμένος να έρθω πίσω, γιατί την 751 που είναι μια θέση σε αποθυματικό που προτείνουν οι πράσινοι το 751 η συγκίτρινη καταπιχη κατά, είναι υπέρ, η πράσινη ε, κατά οι περισσότεροι αποχές απορρίπτεται περνάμε λοιπόν και είμαστε πάντοτε στο Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και εδώ μιλάμε για τεχνική αρρωγή 41-28 Άρτογκ κατά αποχές απορρίπτεται 45-81 ο εισηγητής είναι κατά ποιοι είναι υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται τροπολογία 42 της Επιτροπής Γυναικών η εισηγήτρια είναι κατά ποιοι είναι υπέρ οι σοσιαλιστές όλοι οι άλλοι είναι κατά των γυναικών απορρίπτεται Έχουμε τα σχόλια. Οι τρει επόμενε τροπολογίε έχουν το ίδιο σχόλιο και η συγκήτρια είναι υπέρ. Ποιοι είναι υπέρ, κατά. Αποχές. Αυτές λοιπόν όλες εγκρίνονται. Περνάμε στο επόμενο κεφάλαιο και εδώ έχουμε πολλές ταυτόσιμες τροπολογίες μέχρι το τέλος της σελίδα. Η 354, η συγκίτρια είναι υπέρ, ποιοι είναι υπέρ, κατά. Αποχές δεν υπάρχουν, οπότε εγκρίνονται. Περνάμε στο Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, σε σελίδα 92. Περνάμε στην τροπολογία 41 114. Ποιοι είναι υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 45-20 έχει αποσυρθεί. Έπειτα, οι υπόλοιπε τροπολογίες που, που ακολουθούν είναι θέσεις αποθυματικό και θα τις ψηφίσουμε αργότερα. Περνάμε στη 573 τη Σάλντε, που είναι ταυτόσιμη με τη 4860. Η συγκίτρια είναι κατά. κατά, πολύ, αποχές, μία αποχή. Αυτές οι τροπολογίες απορρίπτονται. Περνάμε στην 715. Η συγγήτρια είναι κατά. Ποιοι είναι υπέρ. Οι σοσιαλιστές. Κατά η πλειοψηφία. Οπότε απορρίπτεται η τροπολογία. Ξαναπάμε πάλι πίσω στην 700. 51 είναι ακόμα μια θέση αποθεματικό που προτείνουν οι πράσινοι. Η συγγήτρια είναι κατά, ποιοι είναι υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. Μετά έχουμε δύο ταυτόσιμες θέσεις σε αποθυματικό. την 761 και τη 4846. Η συγγήτρια είναι κατά, ποιοι είναι υπέρ. Ορισμένοι φιλελεύθεροι. Κατά. Η πλειοψηφία. Αποχές. Απορρίπτονται αυτές οι θέσεις αποθυματικό. Τώρα διαρωτώμε κατά πόσο πρέπει να ψηφίσουμε για τα σχόλια τη 47-62 η εισηγήτρια λέει ναι. Ο κύριος Σούριαν που έχει συντάξει τροπολογία θέλει να ψηφιστεί. Η εισηγήτρια είναι υπέρ αυτή τη τροπολογία. Ποιοι είναι υπέρ. Σας ευχαριστώ. Κατά. Σα ευχαριστώ. αποχέ. εγκρίνεται. Περνάμε στο επόμενο κεφάλαιο. Τροπολογία του κυρίου Άρτονγκ. 41-75. Σας ευχαριστώ υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Η 4521 21 έχει αποσυρθεί. 42-73 Ανδρέασεν υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Η 4522 22 έχει αποσυρθεί. Νομίζω ο κύριος Βαντάλλων έχει αποσύρει όλες. Όχι όλες. 751 θα τη δούμε μετά. Είναι θέση αποθυματικό. Αντίθετα, όλες οι τροπολογίες μέχρι το τέλος της σελίδας είναι ταυτόσιμες. Η συγκήτρια είναι υπέρ, οπότε μ, ψηφίζουμε για την 361. Ποιοι είναι υπέρ, κατά. 360 με συγχωρείτε. Αποχές εγκρίνονται μέχρι κάτω-κάτω στη σελίδα. Οπότε επανέρχομαι στην 751 των πρασίνων. Είναι η ίδια τροπολογία για θέσεις αποθυματικό για τις κλιματικές αλλαγές. Η γήτρα είναι κατά, ποιοι είναι υπέρ. Κατά. Δύο ψηφία, αποχές, δεν υπάρχουν αποχές, απορρίπτεται. Επόμενο κεφάλαιο. Πάντοτε για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερικής Ανάπτυξης. 4176 Άρτογκ υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 45-23 έχει αποσυρθεί. 47-60 έχει αποσυρθεί και αυτή. Και στρέφομαι στον συντάκτη, στον Λάσλο Σούριεν. Λάσλο, έχετε αποσύρει ολόκληρη την τροπολογία ή μόνο τα σχόλια. The whole is withdrawn. Donc, euh, έχει αποσυρθεί. Ωραία, δεν χρειάζεται να ψηφίσουμε. Ψηφίζουμε τώρα για την 362, που είναι ταυτόσιμη με τις τρεις επόμενες. Η ψηγήτρια είναι υπέρ. Ποιοι είναι υπέρ. Σας ευχαριστώ. Κατά. Αποχές εγκρίνονται. Επόμενη σελίδα. Στο επόμενο κεφάλαιο έχουμε τη 4176 του κ. Αρτόγκ. Ποιοι είναι υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται. Έπειτα έχουμε μόνο τροπολογίες για τα σχόλια σε αυτή τη γραμμή. Ψηφίζουμε καταρχήν την 361. Η συγκήτρια είναι υπέρ. Ποια είναι υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 366. Η συγγήτρια είναι υπέρ. Ποιοι είναι υπέρ. Κατά. Η φιλελεύθερη και ο κύριος Άρτογκ. Αποχές. Υπάρχει πλειοψηφία. Υπέρ. Οπότε καλύπτεται και η 536 από αυτήν την ψήφο. Και περνάμε έτσι στην 4759 του κύριου Σούριαν. Που η συγγήτρια είναι υπέρ. Ποιοι είναι υπέρ. Κατά. αποχές εγκρίνεται. Η 4785 καλύπτεται από την 361. Οι παρατηρήσεις δηλαδή της 4785 του κ. Σούριαν καλύπτονται από την ψηφοφορία που έγινε για το 361. Σύμφωνοι, ο κ. Σούριαν είναι ευτυχής, η συγγήτρια επίσης πλέουμε στην ευτυχία, λέει ο πρόεδρος, και αφήνουμε το τέλος της σελίδας που είναι τα πιλωτικά προγράμματα, τα δοκιμαστικά. Η επόμενη σελίδα είναι πάντοτε τα δοκιμαστικά αυτά σχέδια και το άλλο μισό είναι η γραμμή 130331 για τη στρατηγική για την Βαλτική θάλασσα και εδώ Υπάρχουν τρεις τροπολογίες για τις οποίες οι... τα νούμερα έχουν αποσυρθεί. Λοιπόν, τροπολογία 4904. Είμαι υποχρεωμένο να θέσω σε ψηφοφορία τα νούμερα. Διότι ο συντάκτη τη τροπολογία προτείνει να αποσύρει την τροπολογία για τι πληρωμές. Κατάλαβα, αυτό είναι. Ναι, αλλά τότε δεν υπάρχει τροπολογία για τα αριθμού, για τα νούμερα. Ε, Anne, vous pouvez m'expliquer ce que, comment vous comprenez les choses. Uh, Άννα, μπορείτε να μου εξηγήσετε τι συμβαίνει. Η τροπολογία για 2,5 εκατομμύρια στις πληρωμές και τις υποχρεώσεις είναι εντάξει για μας αν είναι 2,5 υποχρεώσεις και 2,5 πληρωμές. Και νομίζω πως η συγγήτρια θα συμφωνήσει με αυτό. Oui, autrement dit, autrement dit, si j'ai bien compris. Δηλαδή με άλλα λόγια αν ε, κατάλαβα καλά, για τις πληρωμές. Στο σχέδιο προϋπολογισμού υπάρχουν 2,5 εκατομμύρια. Δεν υπάρχει αλλαγή, τροπολογία. Αυτό το νούμερο συμφωνείτε, είστε εντάξει. Ωραία. Οπότε, από την άποψη των αριθμών, οι τροπολογίες δεν αφορούν παρά μόνο τις υποχρεώσεις. Εντάξει. Να ψηφίσουμε λοιπόν τα νούμερα και μετά θα ψηφίσουμε και για τα σχόλια. Ωραία. Λοιπόν, για τα νούμερα, το 2,5 εκατομμύρια. Η συγκίτρια είναι υπέρ, ποιοι είναι υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Για τα σχόλια που είναι τα ίδια... Όχι, δεν είναι τα ίδια. Πρέπει να ψηφίσουμε κάθε τροπολογία χωριστά. Α, Υπάρχει συμβιβιστική που λέει να προσθέσουμε τεχνική και διοικητική βοήθεια για το συντονισμό δραστηριοτήτων που σχετίζονται με την Ευρωπαϊκή Στατηγική για την περιοχή της Βαλτικής, χρήματα για το σχεδιασμό και την προετοιμασία προγραμμάτων που στηρίζουν τη στατηγική με τη στήριξη της συμμετοχής της κοινωνίας των πολιτών. Αυτά. Όλοι συμφωνείτε. Α, συνεχίζει να συνεχίζει να βοηθά τις δραστηριότητες των συντονισμού, συμμετέχει στις δραστηριότητες με την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων και αν χρειάζεται από τα βαλτικά κράτη-μέλη στην ανάπτυξη της στρατηγικής για τη Βαλτική Θάλασσα, EU ή e ή κάπως έτσι. Αυτά είναι γραμμένα εδώ. Είναι γραμμένα στο σφακέλο σας. Ναι, Γκέραν. Να διευκρινίσω επίσης ότι αυτό σημαίνει πως το αρχικό κείμενο της Κομισιόν θα διατηρηθεί και ότι η τροπολογία του κύριου Σούριαν ε, στην αρχή έλεγε να διαγραφεί το κείμενο, αλλά συμφωνήσαμε πως όχι και ότι αυτό θα είναι ως προσθήκη στο κείμενο της Κομισιόν. Μάλιστα. Βλέπουμε λοιπόν, ψηφίζουμε αυτό το κείμενο το συμβιβαστικό ως προσθήκη στο κείμενο της Επιτροπής. Σύμφωνοι. Ποιοι είναι υπέρ. Κατά. Αποχές. Δες. Οπότε εγκρίνεται. Και άρα μπορούμε τώρα να ψηφίσουμε για την 4183 του κυρίου Χαρτόγκ. Ποιοι είναι υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Τώρα, προπαρασκευαστική δράση, περνάμε στο, τη σελίδα, γυρίζουμε σελίδα και φτάνουμε στην 99. Λέει ο Πρόεδρος, Ταμείο Συνοχής. Και εδώ έχουμε τρεις ταυτόσιμες τροπολογίες. 3, 63, ο εισηγήτρια είναι υπέρ, ποιοι είναι υπέρ. Ποιοι είναι κατά, αποχές εγκρίνονται. Επόμενο κεφάλαιο, σελίδα 100. Ταμείο συνοχής πάντοτε. 45-24 έχει αποσυρθεί. Οι δύο άλλες, οι επόμενες, αντιστοιχούν σε θέση αποθεματικό. Θα επανέλθουμε σε λίγο. Η πρώτη λοιπόν που θα ψηφίσουμε είναι η 42-74 της κυρίας Ανδρέασεν. Ποιοι είναι υπέρ. 2 κατά. Σας ευχαριστώ. Αποχές απορρίπτεται. Η 751 είναι πάλι θέση σε αποθεματικό των πρασίνων. Θα επανέλθουμε. Ψηφίζουμε για τη 10-19 της Γκουε. Η συγκίτρινη κατά. Ποιοι είναι υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 574. Η συγκίτρινη υπέρ. Ποιοι είναι υπέρ. κατά αποχές όχι συγγνώμη συγγνώμη έκανα λάθος η συγκίτρια ήταν κατά ναι, ναι. Όταν πρόκειται για τους φιλελεύθερους είναι η καρδιά μου που μιλάει. Κοιτώ την Άννα. Με συγχωρείτε. Λοιπόν, η 4861 έχει απορριφθεί και αυτή και η 574 γιατί ήταν ταυτόσιμε. Τώρα ψηφίζουμε για την 716 που η συγκήτρια είναι υπέρ. Ποιοι είναι υπέρ. Οι σοσιαλιστέ μάλιστα. Ποιοι είναι κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Πάμε πίσω στην 562. θέση αποθυματικό. Που είναι ίδια με την επόμενη. Αλλά η συγκήτρια δεν τη θέλει υπέρ, ποιοι είναι κατά αποχές. Αυτές οι δύο τροπολογίες απορρίπτονται. Και ψηφίζουμε την 751 των Πρασίνων για τις κλιματικές αλλαγές. Φαντάζομαι την ίδια πλειοψηφία. Ποιοι είναι υπέρ, οι πράσινοι φίλοι μας, κατά. Απορρίπτεται και εδώ. Έρχομαι κάτω-κάτω στην ίδια σελίδα που έχουμε να ψηφίσουμε τα σχόλια. 536 είναι η τροπολογία. Η συγκεντρία είναι υπέρ. Ποιοι είναι υπέρ. Σας ευχαριστώ. Κατά. Ας κάνουμε μία ε, ηλεκτρονική επαλήθευση για να ξυπνήσουμε κιόλας. Ψηφίζουμε. Συμμετέχω κι εγώ στην ψηφοφορία, εκτός αν κάποιος μου πει όχι. Ψηφίζουμε. Δύο κάρτες είναι στη θέση τους, αλλά δεν έχετε ψηφίσει. Τέλος της ψηφοφορίας. 15 υπέρ, 22 κατά, απορρίπτεται. Γι' αυτό πρέπει να ψηφίσουμε για την 367. Όχι, είναι ταυτόσιμη. Ε, απορρίπτεται και αυτή λοιπόν. Μάλιστα, περνάμε στην ε, διασυνοριακή συνεργασία. 41-85 Αρτόγκ. Η εισηγήτρια είναι κατά, ποιοι είναι υπέρ. Ο κύριος Άρτογκ. Ποιοι είναι κατά. Η πλειοψηφία, πολύ εχθρική, αποχές απορρίπτεται. 168 της ε, ΑΦΕΤ δεν τη θέλει η εισηγήτρια. Ποιοι είναι υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. Πολύ ωραία. Χαρακτηρία στην εισηγήτρια. 40% του προπολογισμού ήδη έχει περάσει. Δεν είναι και άσχημα. Περνάμε λοιπόν τώρα στην κατηγορία 2. Γεωργία. Euh, l'amendement 67, le rapporteur est pour. Qui est pour? Τροπολογία 67. Η συγκίτρια είναι υπέρ. Ποιοι είναι υπέρ? Έχετε όλοι τον κατάλογο. Υπέρ, κατά, αποχές. Εγκρίνεται. Δεν σηκώσατε και πολύ τα χέρια, πάντως τα πιο πολλά χέρια ήταν υπέρ. Εγκρίνονται αυτές τις τρεις λοιπόν. Στην επόμενη σειρά, γραμμή. 41-38 Κατά, Κατά παχές απορρίπτεται. Η 68 υπέρ. Ο εισηγητής είναι υπέρ. Ευχαριστώ. Κατά αποχές εγκρίνεται και καλύπτει τις δύο επόμενες τροπολογίες που είναι ταυτόσιμες. Γυρίζω τη σελίδα 102 πάνω στη σελίδα είναι ένα πιλωτικό πρόγραμμα. 996 ε, που είναι η ταυτόσημη 499. Ο εισήγης είναι κατά ποιος είναι υπέρ. Κατά. Θα κάνουμε μια ηλεκτρονική επαλήθευση. 996 και 499 άρχεται ψηφοφορία. Ψηφίστε λοιπόν. Υπάρχει ένα σοσιαλιστής παραπάνω. Παρακαλείτε να αποσυρθεί. Πέραση της ψηφοφορίας. Εφτά υπέρ, 30 κατά. Δεν καταλαβαίνω τίποτα. Άρα απορρίπτεται. Δεν ήταν καθαρό από τη δική μου προπτική το αποτέλεσμα. Φαίνεται ότι κάποιοι είναι κουρασμένοι. Είναι η ώρα της σιέστας στις μεσογειακές χώρες. Θα περάσουμε στα προγράμματα υπέρ των απόρων. 42-66, ε, ο είναι κατά υπέρ. Κατά αποχές Κανείς δεν είναι υπέρ, ούτε στην ομάδα των ε, συντακτών. υπέρ. Ο συντάκτης κατά. Δυστυχώς μια πλειοψηφία εποχές απορρίπτεται λοιπόν. Στη συνέχεια θα υποβληθεί η 803 πριν από την 97 γιατί είναι αυτή η οποία απομακρύνεται περισσότερα. 803, ο σύγκτης είναι υπέρ. Ποιος άλλος είναι υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Καλύπτει όλες τις άλλες μέχρι το τέλος της σελίδας. Αλλά θα πρέπει να επανέλθω στο σχόλια. Α, λέει ο πρόεδρος, δεν χρειάζεται να το ξαναφέρουμε, είναι αποκλειστικά πρόκειται για σχόλια, αλλά περνάμε στην επόμενη σελίδα 103 και έχουμε την 69 υπέρ, ο συγητής υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 997 της γκουε, ο είναι κατά, υπέρ. κατά αποχές απορρίπτεται. Η 598η, άρα απορρίπτεται ταυτόσημη άρα απορρίπτεται. Η 98 να μπει στο αποθηματικό. Ο εισηγητής είναι υπέρ. Υπέρ παρακαλώ. Κατά η φιλελεύθερη και ο κύριος Αρτόγκ. Αποχές Εγκρίνεται λοιπόν να μπει στο αποθεματικό η 70. Ο εισηγητής είναι υπέρ. Ποιο άλλο είναι υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Στη συνέχεια κύριε Σιγητά, με συμβουλεύουν να ε, υποβληθεί τη ψηφοφορία καταρχήν η 71 που είναι στην επόμενη σελίδα. Η 71 που είναι στην αρχή της σελίδας 119 στο ελληνικό κείμενο. με έναν, αριθμό 205 εκατομμύρια υποχρεώσεις. Και πληρωμές επίσης, λέει ο Πρόεδρος. Συμφωνείτε? Άρα λοιπόν είναι η 71 Βρισκόμαστε στη γραμμή κατά μία οργανώσεων παραγωγών. Η τροπολογία που έχει προταθεί από τον εισηγητή αφορά 205 εκατομμύρια. Το καταλάβατε όλοι. Ωραία. Υπέρ. Ευχαριστώ. Κατά. Η φιλελεύθερη και ο κύριος Αρτόγκ. Αποχές. Ωραία. Ευχαριστώ. Εγκρίνεται. άρα καλύπτει τη 47-27, Θα πρέπει λοιπόν να ψηφίσουμε την 72. Συγγνώμη, λέει ο πρόεδρος. Υπάρχουν κάποιες παρατηρήσεις, άρα θα πάμε πίσω

Συγγνώμη, λέει ο πρόεδρο. ε, μου έδωσαν ε, συμβουλέ. Η 92 και η 93. Πρόκειται για την 92 μάλλον και την 93. Λοιπόν, όχι. Τις αφήνουμε. Λοιπόν, ε, ε, θα Ε, θα ξαναψηφίσουμε το 255 εκατομμύρια. Ο Τζοβάνι Λαβίο Βία έχει το λόγο. Κοιτάξτε, σε αυτά που μας δώσατε γίνεται λόγος για αύξηση 70, ε, κατά 75, ενώ εδώ είναι 175. Ε, λοιπόν, αυτό είναι το νούμερο. Σωστό είναι. Λοιπόν, με άλλα λόγια, τα σχόλια για αυτό την τροπολογία 71, υπαριθμόν 71, η Επιτροπή θα παρουσιάσει μια πλήρη πρόταση στο Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο για να εξασφαλίσει ότι η αύξηση 175 εκατομμύριων κλπ. κλπ. θα χρησιμοποιηθεί, είναι χρήσιμη κλπ. κλπ. Έχετε αυτό το κείμενο μπροστά σας. Ποιος είναι υπέρ αυτού του σχολείου. Κατά αποχές οι πράσινοι απέχουν. Εγκρίνεται συνεπώς. Άρα λοιπόν δεν έχουμε ανάγκη να πάμε προς τα πίσω να ξαναγυρίσουμε πίσω. Το 72, η 72, συγγνώμη, ε, υποβάλλεται σε ψηφοφορία, 72, με ποιο νούμερο. 95 εκατομμύρια μου λένε. Αυτό είναι το νούμερο. Ωραία, ωραία. όχι 20 εκατομμύρια, αλλά 95 Ωραία λοιπόν. Η τροπολογία υπαριθμών 72 και πρόκειται για 95 εκατομμύρια υπέρ. Κατά. Ευχαριστώ. Αποχές. Εγκρίνεται. Και στη γραμμή αυτή επίσης έχουμε, χρειαζόμαστε τα ίδια σχόλια τα οποία ψηφίσαμε για την 71 αλλά με ένα διαφορετικό νούμερο που αυτή τη φορά είναι 75. Ωραία λοιπόν. Υπέρ. Υποθέτω η ίδια πλειοψηφία. Πρόκειται για το ίδιο πράγμα στην ουσία. Κατά. Αποχές. Άρα εγκρίνεται επίσης. Άρα λοιπόν εγκρίναμε 250 ε, εκατομμύρια από τη μία και 95 από την άλλη με τα ίδια σχόλια. δηλαδή ζητούμε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να εξασφαλίσει ό,τι κλπ. κλπ. Ωραία λοιπόν. Τώρα θα περάσουμε στη διανομή των φρούτων στα σχολεία. 73. Ο Σίγης είναι υπέρ. Ποιος άλλος είναι υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται και καλύπτει όλη τη σελίδα αυτή. Στην επόμενη σελίδα επάνω ε, 41-39 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 74 της Επιτροπής Γεωργίας Συστής είναι υπέρ. υπέρ. Ευχαριστώ. Κατά αποχές εγκρίνεται καθώς και οι ταυτόσιμες τροπολογίες στην ίδια γραμμή. Θα περάσουμε λοιπόν στα λοιπά μέτρα για τον αμπελονικό τομέα. Υπέρ, ο κύριος Σαρτόγκ. Συγγνώμη, λέει ο πρόεδρος. Κατά, αποχές απορρίπτεται. 75 της υπέρ, ο σύγκτης είναι υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Ενέργειες πρόθεσης 76, ο εισηγητής είναι υπέρ, υπέρ παρακαλώ. Κατά. Ευχαριστώ, αποχές εγκρίνεται. Στη συνέχεια έχουμε την 93 ο εισηγητής είναι υπέρ. Υπέρ παρακαλώ. Ευχαριστώ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Πιλωτικό σχέδιο για το γάλα. 998. Ο κατά. Υπέρ. Ευχαριστώ. Κατά αποχές απορρίπτεται. Στο γάλα στα σχολεία, 41-41, υπέρ. Κατά, αποχές, απορρίπτεται. 91 της Επιτροπής Γεωργίας, υπέρ. Κατά, αποχές εγκρίνεται καθώς και οι τροπολογίες που καλύπτονται μέχρι το τέλος της σελίδας και τώρα θα περάσουμε σε επιστροφές στο βόλιο Κρέας 999. ποιος είναι υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται το ίδιο και επόμενε. 77. Ε, ο είναι υπέρ. Ποιος είναι κατά. Αποχές εγκρίνεται. Επιστροφές τη ζώντα ζώα. Χίλια. Υπαριθμόν χίλια. Ο είναι κατά. Υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. Η 503 καταπίπτει χείριο κρέας. 1001. Ο είναι κατά. Υπέρ. Κατά. Κατά του χείριου κρέαστος απορρίπτεται. 504 καταπίπτει. Αυγά. 1002. Ο Σύρης είναι κατά. Ποιος είναι υπέρ των αυγών. 5. Κατά των αυγών. Ευχαριστώ. Έγινε ο μελέτα και οι δύο τροπολογίες απορρίπτενται. Η 78 εισηγητής είναι υπέρ για τα αυγά πάλι. Κατά αποχές η 78 εγκρίνεται συνεπώς. Και τώρα θα περάσουμε στο κρέας πουλερικών. Η 1003 ο εισηγητής είναι κατά, υπέρ. Ευχαριστώ κατά αποχές απορρίπτεται, καθώς και 505. Στη συνέχεια έχουμε πιλωτικό σχέδιο. Ε, καπνός. 622 των φιλελευθέρων συγκητής είναι υπέρ. Ποιος άλλος είναι υπέρ. Κατά. Το ΕΛΚ. Αλλά είναι απομονωμένο. Α, όχι. Υπάρχουν και σοσιαλιστές που καπνίζουν. Μάλιστα. Ωραία, λοιπόν. Ηλεκτρονική επαλήθευση. Άρχεται η ψηφοφορία. Ευχαριστώ οι φίλοι του καπνού και οι φίλοι του καρκίνου, πέρας της ψηφοφορίας. 17 υπέρ, 19 κατά, απορρίπτεται. Το 2004 τώρα, όχι, είναι ταυτόσιμος. Όχι, καταπίπτουν όλες. Ε, 48-12. Ο εισηγητής είναι κατά. Ποιος είναι υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. Τώρα το 41-42, όχι είναι ταυτόσιμο του κυρίου Χαρτόγκ, άρα καταπίπτει. Τίποτα δεν γίνεται με τον καπνό. Τέλος ο καπνός, το κάπνισμα. Λοιπόν, αποχή των καπνιστών. Λοιπόν, 79. Ο εισηγητή είναι υπέρ. Ποιο άλλο είναι υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Η ενίσχυση της 41 41-43 του κ. Αρτόγκ υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται. Βαμβάκι 80 εισηγητής είναι υπέρ. υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Οι συνδεδεμένες άμεσες ενισχύσεις 81, ο συγκριτής είναι υπέρ, Κατά αποχές εγκρίνεται. 82, η συγκριτής είναι υπέρ. Υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Η 512. Προπαρασκευαστική δράση. Ο εισηγητής είναι κατά. Υπέρ παρακαλώ. Η πράσινη. Κατά. Όλοι οι άλλοι αποχές, αλλά απορρίπτεται. Αντιθέτως θα πρέπει να ψηφίσουμε το, τα σχόλια για το 45-25 ο εισηγητής είναι κατά. Α, όχι, είναι υπέρ. Υπέρ ο εισηγητής. Υπέρ. 45-25. Κατά. Αποχές. Άρα το, σχόλιο, ε, το σχόλιο δεν, είναι, δεν θα πρέπει να χρησιμοποιείται για τη τεχνολογία της κλωνοποίησης. Απορρίπτεται. Τώρα, προγράμματα αγροτικής ανάπτυξης 83 της Γεωργίας. Ο εισηγητής είναι υπέρ. Υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Καθώς και όλες οι ταυτόσιμες τροπολογίες που ακολουθούν σε αυτή τη γραμμή. Στο επόμενο κεφάλαιο, επιχειρησιακή τεχνική βοήθεια. 45-90. Υπέρ. Ο εισηγητής είναι κατά. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. Η 84. Ο εισηγητής είναι υπέρ. Υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Τώρα γυρνάω τη σελίδα πιλωτικό σχέδιο, πιλωτικό πρόγραμμα, ε, καθάριση των λογαριασμών. Η 87 υπέρ κατά ευχαριστώ εγκρίνεται. Έρευνες για τη διάθεση των γεωργικών εκμεταλλεύσεων 41-45. Υπέρ. 2. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 88. Της Επιτροπής Γεωργίας Συστήγης είναι υπέρ. Υπέρ. Ευχαριστώ. Κατά. Εγκρίνεται. 41-46 του κυρίου Αχατόγκ. Υπέρ κυριος Άρτονγκ. Κατά αποχές απορρίπτεται. 41-47 του κυρίου Άρτονγκ. Υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται. 851 το συντηρητικό Ο είναι κατά. Υπέρ. 4. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. Και η επόμενη. 89. Γεωργία. Υπέρ ο συγκριτής. Υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 90 της Επιτροπής Γεωργίας, υπέρ, υπέρ. Ευχαριστώ κατά αποχές εγκρίνεται. Στη συνέχεια έχουμε τα πιλωτικά προγράμματα. Στη μέση της σελίδας, στη γραμμή live, 41-51 του κ. Χαρτόγκ, υπέρ κατά, αποχές απορρίπτεται. 479 τη Επιτροπής Περιβάλλοντος υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. Η επόμενη γραμμή, 4153 του κ. Αρτόγκ υπέρ, κατά, αποχές απορρίπτεται. 477 που υποστηρίζεται από τον εισηγητή. Υπέρ, παρακαλώ. Κατά, αποχές εγκρίνεται. Η επόμενη γραμμή, επίσης το live, 4155 του κυρίου Αρτόγκ, υπέρ, κατά, απορρίπτεται. 854 των συντηρητικών, υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 478 της Επιτροπής Περιβάλλοντος, της είναι υπέρ, υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Το ίδιο και όλες οι ταυτόσιμες τροπολογίες μέχρι το τέλος της σελίδας. Περνάμε τώρα στην επόμενη σελίδα στον οργανισμό περιβάλλοντος. 4156 του κ. Χάρτονγκ. Υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. Η 4526 έχει αποσυρθεί. 1 με τη συμφωνία του εισηγητή υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται καθώς και οι επόμενες τροπολογίες που είναι ταυτόσιμες στην ίδια γραμμή. Θα περάσουμε στη συνέχεια σε μια άλλη γραμμή πάλι για τον οργανισμό περιβάλλοντος, συνεισφορά στον τίτλο 3, 4157 του κ. Χάρτο Μεσητής είναι κατά. Ποιος είναι υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται. Η 4527 έχει αποσυρθεί. Στη συνέχεια έχουμε πλωτικά προγράμματα ε, και επόμενες σελίδες. Φτάνουμε στον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Χημικών. 470. Ποιος είναι υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Η επόμενη γραμμή του Βαντάλεν έχει αποσυρθεί. 469. Ε, Ποιος είναι υπέρ. Ευχαριστώ κατά. Ευχαριστώ αποχές. Εγκρίνεται. Η 4531 έχει αποσυρθεί. Ένα νέο ε, πιλωτικό πρόγραμμα και φτάνουμε στην τροπολογία του κυρίου Χάρτογκ 4163 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 911 ο συγητής είναι κατά. Ποιος είναι υπέρ Αποχές απορρίπτεται. 46... Η 46-25 ε, υπέρ κατά απορρίπτεται. Είμαστε στη σελίδα 142 του ελληνικού κειμένου. Θα περάσω στην Αλία λοιπόν. 105 ε, υπέρ κατά 115 συγγνώμη εγκρίνεται καλύπτεται και επόμενη του πόρτας λοιπόν 10-16 σελίδα 143 υπέρ παρακαλώ κατά αποχές ομοφωνία κατά απορρίπτεται γερνάω τη σελίδα Είμαστε στα προγράμματα αλίας για τις περιφερειακές περιοχές του κυρίου Αρτόγκ. Υπέρ κατά απορρίπτεται. 10-17 της Γκουε. Ο εισηγητής είναι κατά. Ποιος είναι υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Και η επόμενη καταπίπτη. Στη συνέχεια έχουμε τα πιλωτικά προγράμματα Διεθνής Συμφωνίας για την Αλία ε, του κυρίου Αρτόγκ. 42 63 σχόλια. Ο εισηγητής είναι κατά. Ποιος είναι υπέρ αυτών των σχολείων. Ευχαριστώ. Αποχές. Πρόκειται με περίεργη πολιτική γεωμετρία. Αλλά νομίζω ότι απορρίπτεται τελικά η τροπολογία. 128. Ο εισηγητής είναι υπέρ. Ποιος άλλος είναι υπέρ. Κατά. Ευχαριστώ. Εγκρίνεται. Η επόμενη γραμμή. 4171 του κυρίου Χάρτογκ. Υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 122 Επιτροπή Αλίας υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Η επόμενη ταυτόσημη επίσης απορρίπτεται. Περνάμε στο Ευρωπαϊκό Ταμείο Αλίας. 856 των συντηρητικών. Ο είναι κατά. Υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. Η 123 της Επιτροπής Αλίας υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται και όλες στις μεστροπολογίες που ακολουθούν στην διαγραμμή του προπολογισμού. Στη συνέχεια έχουμε κάποια πιλωτικά προγράμματα. Λοιπόν, και έρχομαι αμέσως στη μέση της σελίδας 4172 του κυρίου Χάρτονγκ υπέρ κατά Αποχές απορρίπτεται. 857 το συντηρητικών ασχεδίων είναι κατά υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. Η 116. Υποστηρίζει ο εισηγητής υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Θα περάσουμε τώρα στην επόμενη γραμμή 4172 του κυρίου Χάρτον. υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. Η 1018 της Γκουε υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται το ίδιο και η επόμενη 117 του Σιγητού υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται ε, πιλωτικά σχέδια ε, συνεχίζει η επόμενη σελίδα και φτάνουμε στην 118 που υποστηρίζει ο εισηγητής. Είναι υπέρ της 118. Υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Ο εισηγητής συνεχίζει να σηκώνει το χέρι. Ε, ήταν υπέρ της 118. Λοιπόν, περνάμε στην κοινοτική υπηρεσία ελέγχου της Αλίας. 45-32 έχει αποσυρθεί. Η 120 έχει την υποστήριξη του, του υπέρ παρακαλώ για την 120 κατά. Ευχαριστώ αποχές. Εγκρίνεται. Και η τροπολογία της κυρίας Χάου καλύπτεται. Θα περάσουμε στη 45-32 έχει αποσυρθεί. Στην 119 της Επιτροπής Αλίας. Υπέρ παρακαλώ. είναι υπέρ. Ευχαριστώ κατά. Αποχές εγκρίνεται. καλύπτεται της Γιούτα. Ε, η 353, συγγνώμη λέει ο πρόεδρος, ναι, για την πρωτοβουλία πολιτών, 353. Θα έπρεπε να είναι στην κατηγορία 3 μου λένε. 3β. Μπορούμε να την ψηφίσουμε και μετά αν εγκριθεί να τη βάλουμε στην 3β. Άρα ο εισηγητής είναι υπέρ υπέρ των πολιτών, κατά των πολιτών, εγκρίνεται αποχές. Εγκρίνεται, λοιπόν, θα τη βάλουμε, όπως είπαμε, στο 3β. Ωραία, λοιπόν. Θα περάσουμε στον εκτελεστικό οργανισμό για την υγεία και τους καταναλωτές. Η μόνη τοπολογία δεν έχει αποσυρθεί. Στη συνέχεια έχουμε πιλωτικά προγράμματα στα μέσα της σελίδας για τις ασθένειες των ζώων που ενδιαφέρουν την ΚΟΕ. 975 που υποστηρίζει ο εισηγητής. Ποιος είναι υπέρ. Κατά των ασθενειών των ζώων. Αποχές. Τα ζώα σώθηκαν λοιπόν. Ε, πάλι έχουμε προγράμματα πιλωτικά. Οι 57, ακόμα, συνεχίζουμε να είμαστε στα ζώα. 57, ο συγκεκριτής είναι υπέρ. Ποιος άλλος είναι υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Επίσης όλες οι επόμενες απολογίες που είναι ταυτόσιμες. Στη συνέχεια έχουμε τη 4682 που πρόκειται για τις φυτογενομικές παρεμβάσεις. Μου λένε ότι η συγκτής είναι κατά ε, της τροπολογίας για το νούμερο, αλλά είναι υπέρ του σχολείου. Καταρχήν να ψήσουμε για το νούμερο. Ο εισηγητής είναι κατά. Ποιος είναι υπέρ ουδής. απορρίπτεται. το σχόλιο, συγητής είναι υπέρ. Ποιος είναι υπέρ. Ηλεκτρονική επαλήθευση. Άρχεται η ψηφοφορία. Όλο και περισσότερο ψηφίζουμε. Τέλος της ψηφοφορίας. 14 υπέρ 25 κατέ. Τα έχουμε τα πρότυπα σχέδια, τα πιλωτικά και έτσι τελειώνουμε την κατηγορία 2. Τώρα να διανύμουμε το κατάλογο ψηφοφορίας για την κατηγορία 3. Φραντσέσκα. Στρέφουμε στην ησυχήτρια για την κατηγορία 3α. Υπάρχουν νέα στοιχεία σε σχέση με αυτά που είχαμε προετοιμάσει. Έγιναν συζητήσεις στη διάρκεια του μεσημεριανού. Αλλαγές υπάρχουν που πρέπει να ξέρουμε πριν να ψηφίσουμε. Εγώ θα έλεγα ότι μπορούμε να ψηφίσουμε τώρα, ναι, στο αυτό το νέο, τη νέα κατηγορία. Λοιπόν, με βάση λοιπόν τον πίνακα συνεχίζουμε με την 977. είναι το Ευρωπαϊκό Ταμείο για τους Πρόσφυγες. Υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 100 εκατομμύρια. 978 της ΓΚΟΕ. Η εισηγήτρια είναι κατά, ποιοι είναι υπέρ. Κατά, αποχές, απορρίπτεται. Η 4708 επίσης. Πρέπει να ψηφίσουμε τη 4708. 08 ε. Bon, de toute façon, est-ce Κάποιο το υπερασπίζεται αυτό. Οι συντάκτε δεν είναι εδώ. Κανένα δεν είναι εδώ. Λοιπόν, αντίο σα. Την περνάμε suivante, en haut 979 η υπέρ, ποιοι είναι υπέρ, κατά. Αποχές εγκρίνεται. Και οι δύο υπόλοιπες. Ευρωπαϊκό Ταμείο Επιστροφών. 1061. Η είναι κατά, ποιοι είναι υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. Και άρα καταπίπτει και η 10 Δέκα 60 της Γκουε. Η συγκίτρινη κατάπιν υπέρ. Κύριε κυρία Ανδρέασεν και ο κύριος Χάρτογκ. Κατά αποχές. Απορρίπτεται. Και η 4710. 430 λίμπε υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Στην επόμενη γραμμή, Ευρωπαϊκός Οργανισμός για τη διαχείριση της επιχειρησιακής συνεργασίας στα εξωτερικά σύνορα. Η Frontex δεν είναι αυτή, ναι. Λοιπόν, ο Βαντάλεν έχει αποσυρθεί. Ψηφίζουμε πρώτα για τα νούμερα από την 444 και κάτω. Ποιοι είναι υπέρ, κατά, Κατά των νούμερων αυτών, ε, αποχές, η πλειοψηφία είναι υπέρ. Ωραία. Για αυτή τη γραμμή δεν υπάρχει άλλη τροπολογία. Πρέπει να ψηφίσουμε την 927. Α, καλύπτεται. Ωραία λοιπόν, για τα νούμερα ξεκαθάρισε το τοπίο, τώρα όμως πρέπει να ψηφίσουμε για τα σχόλια. Τα σχόλια του 444. Η θηγήτρια είναι υπέρ. Ποιοι είναι υπέρ. Κατά. Αποχές. Πλειοψηφία για τα σχόλια. Λοιπόν, θεωρούμε ότι ε, και οι δυο άλλες τροπολογίες καλύπτονται. Όχι, πρέπει να τις ψηφίσουμε και αυτές. Πρέπει να ψηφίσουμε τα σχόλια για την 752. Είναι συμβατό. Μπορεί να προσθεθεί. Η εισηγήτρια συμφωνεί. 752 σχόλια. Α, όχι. Η εισηγήτρια είναι κατά. The remarks, the remarks. Now I know who is controlling you. Yeah, yeah. Madame, Madame le rapporteur, dites-moi. Για μπείτε μας κυρία εισηγήτρια. Λοιπόν, για την 752 οι παρατηρήσεις είναι συμβατές και η πρότασή μου είναι υπέρ. Εγώ είμαι υπέρ. Donc, du 752. Le Η εισηγήτρια λοιπόν είναι υπέρ. Ποιοι είναι υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 753. Οι παρατηρήσεις είναι συμβατές. Ναι, και εσείς είστε υπέρ. Ωραία. Υπέρ, κατά, αποχές. Εγκρίνεται. Όλες λοιπόν αυτές οι παρατηρήσεις εγκρίνονται, είναι συμβατές. Πάμε παρακάτω. Οι 44-62 είχε αποσυρθεί, οι δύο επόμενες είναι ε, αποθεματικά και σχόλια, θα επανέλθουμε και ψηφίζουμε για την 9-28 ποιοι είναι υπέρ. και είναι υπέρ της 928. Η συγγήτρια, η ομάδα σας έχει πάθει σύγχυση. Και νομίζω ότι θα ήθελαν να ψηφίσουμε πρώτα τα νούμερα. Τις 459. Ε, πείτε μου τι να κάνουμε. Ε, Possiamo votare prima anche i 400... Μπορούμε να ψηφίσουμε πρώτα την 459 και την 754 μετά με τα νούμερα που είναι συμβατές, κατά τη γνώμη μου. Μάλιστα, θα ψηφίσουμε λοιπόν θα ψηφίσουμε λοιπόν 459 και την 754 που είναι τα ίδια τα νούμερα και θα επανέλθω μετά σε αυτές τις τροπολογίες όσον αφορά τα σχόλια και τη θέση θεματικό. Λοιπόν, νούμερα 25 εκατομμύρια. Ποιοι είναι υπέρ μαζί με την εισηγητρία. Κατά. Κατά. Αποχές. Πλειοψηφία είναι υπέρ. Και τώρα λοιπόν πάμε στις επόμενες 9.28, 45.61 και 43.89 οι οποίες καλύπτονται από τους αριθμούς που μόλις ψηφίσαμε. Επανέρχομαι λοιπόν σε αυτές τις δύο τροπολογίες για να ψηφίσουμε καταρχήν την θέση αποθεματικό. Τα σχόλια θα ψηφίσουμε, τα σχόλια. Λοιπόν, τα σχόλια της 459. Η εισηγήτρια είναι υπέρ. Ποιοι είναι υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνονται τα σχόλια. Σχόλια τώρα του 754. Καλύπτεται, καλύπτεται. Άρα δεν χρειάζεται να ξαναψηφίσουμε. Ωραία. Ωραία λοιπόν. Όλα είναι ξεκάθαρα για αυτή τη γραμμή διαφορετική ψήφος από αυτή που πρότεινε η συγκίτρια, αλλά, εν πάση περιπτώσει, τέλος τώρα εδώ. Τελειώσαμε. Και περνάμε στο Σέγγεν. ΣΥΣ 2. Έχουμε θέσει αποθυματικό. 4.45 και 7.55. Η συγκίτρια είναι υπέρ. Ποιοι είναι υπέρ? Κατά. Αποχές. Εγκρίνονται. Visa λοιπόν, η είναι υπέρ. Άλλη υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Ερχόμαστε τώρα στο Ταμείο Εξωτερικών Συνόρων. 460. Η είναι υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Donc ça couvre les Καλύπτει τα επόμενα τρία και η τροπολογία τώρα 731. Ψηφίζουμε απλώ τα σχόλια. Η συγκήτρια υπέρ, άλλο υπέρ. Κατά. απόχέ. εγκρίνεται. Εξελόγηση Σέγγεν. Για να εγγραφεί το αποθεματικό ρώταση η υπέρ, άλλη υπέρ. Κατά. απόχέ, εγκρίνεται. Je tourne la page. Γυρνάω σελίδα. Ευρωπαϊκό Ταμείο Επιστροφής. 1059 της ΓΚΟΕ εισηγήτρια. Κατά. Και Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Όπως και η επόμενη λοιπόν. 361. Ε, Πρώτα τα ποσά και μετά τα σχόλια θα δούμε. Η εισηγήτρια είναι υπέρ. Ψήφι υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Donc ça couvre les deux amendements ε, επόμενα, λοιπόν, καλύπτω το 858. Η συγκήτρια είναι κατά. Άλλη υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίψετε. Άρα, επανέρχομαι στα σχόλια της 461. Η συγκήτρια είναι υπέρ. Ψήφι υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Je reviens alors au 732. Επανέρχομαι στο 732. Ε, fundamental rights. Ε, τα σχόλια συγκεκριμένων υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται για τα θεμελιώδη δικαιώματα. Επόμενο κονδύλι έχει αποσυρθεί η τροπολογία όπως και η μεθεπόμενη. Πάμε στην επόμενη σελίδα ψήφι παίρνει για το Ταμείο της Πρόσφυγης. Κατά αποχές απορρίπτεται. Του κυρίου Χάρτον και 4205. 729. Η είναι υπέρ. Ψήφι υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Λοιπόν, στην 447... Και εφόσον έχει εγκριθεί 729, αφορά μόνο την ανάληψη υποχρεώσεων. Τη θέτω λοιπόν σε ψηφοφορία μόνο για τις πληρωμές, διότι για την ανάληψη υποχρεώσεων έχει εγκριθεί. Καλύπτεται από την προηγούμενη που ψηφίστηκε. Ah, pardon. Le secrétariat fait μου επισημαίνει και σωστά η γραμματεία ότι για τις πληρωμές, η τροπολογία που απέχει περισσότερο είναι η 1058. Οπότε θα πρέπει να ψηφίσουμε πρώτα αυτή που ταυτίζεται με το 4713 πριν την 447. Μόνο τις πληρωμές ψηφίζουμε. Για την ανάληψη υποχρεώσεων έχουμε αποφασίσει. Γιατί εγκρίναμε την προηγούμενη και είναι 20 εκατομμύρια στην 729. Λοιπόν, αυτό που ψηφίζουμε τώρα αφορά μόνο τις πληρωμές. Και για τις πληρωμές το μεγαλύτερο ποσό είναι η τροπολογία 1058. Και η συγκίτρια είναι υπέρ. Είναι γενναιόδωρο το κοινοβούλιο στις πληρωμές. Ψήφι υπέρ μαζί με την εισηγήτρια. Κατά. Αποχές. Άρα λοιπόν οι 10.58 και 47.13 εγκρίνονται σε ό,τι αφορά τις πληρωμές, ενώ τα υπόλοιπα καταπίπτουν. Και σε αυτό το κονδύλι έχουμε ακόμα τα σχόλια της Επιτροπής Προπολογισμών σε ό,τι αφορά τις γυναίκες. Είναι του Σούριαν η τροπολογία. Ψήφι υπέρ μαζί με την ισχύτρια κατά. Α, όχι, όχι, ισχύτρια κατά. Ζητώ συγγνώμη. Λοιπόν, ε, τότε ηλεκτρονικά να το λέξουμε προτιμώ. Για τα σχόλια της τροπολογίας 4764 αυτό που προτείνει για τις γυναίκες ο Λάσλο Σούριαν. Sorry, αλλά... Uh, Άρχεται η ψηφοφορία. Ah, thank you. Thank you. very much. Le vote est ouvert sur les femmes. Άρχεται η ψηφοφορία για τις γυναίκες. Le vote est clos. Le vote est clos. Le vote est clos. Πέρας. 16 pour. 21 υπέρ, 21 μέλη της Επιτροπής Προϋπολογισμών δεν συμφωνούν με το όραμα του Λάσλο Σούρλια για τις γυναίκες. Άκουσαν, άκουσαν. Και τα σχόλια απορρίπτονται. Λασλό, encore du lobbying à faire. Α, εδώ έχει πολλή δουλειά ακόμα για λόμπι. Πάμε παρακάτω. Έκτακτα μέτρα σε περίπτωση μαζικής εισρωής προσφύγων. 730 εδώ ξαναπέφτουμε σε μια σειρά τροπολογιών που έχουμε και ανάληψη υποχρεώσεων και πληρωμε 7.30. Η συγκήτρια είναι υπέρ της ανάληψης υποχρεώσεων. Άλλη υπέρ. Κατά. Αποχές. 200 εκατομμύρια εγκρίνεται. Όχι, 200.000 διορθώνει ο πρόεδρος. Ε, δεν είναι και πολλά λεφτά αυτά. Le secrétariat a décidé qu'il y avait 3-0 de moins. Bon, bon d'accord. Très bien. Alors... Λοιπόν, συνεχίζουμε. Πληρωμέ τώρα. Έχει μεγάλη πλάκα εδώ. Γιατί έχουμε 200.000 ανάληψη υποχρέωσεων και 2,5 εκατομμύρια πληρωμέ. Να δω πώ θα τα βγάλουμε πέρα. Ε, λοιπόν, πληρωμέ. Τρει ταυτόσιμε τροπολογίε. Η συγκίτρια είναι υπέρ. Άλλο υπέρ. Κατά. Merci, attention. Αποχές. Υπάρχει μια πλειοψηφία λοιπόν υπέρ. Άρα θα μειωθεί το υπόλοιπο προς εκαθάριση, το περίφημο ραλ. Πολύ αριθμητική είναι. Όχι, είναι πολύ ειδική, μόνο εμείς τα καταλαβαίνουμε. Εν πάση περιπτώσει, οι πολίτες θα ε, μείνουν ικανοποιημένοι. Συνεχίζουμε. 42.06 χάρτων. Ψήφι υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Η επόμενη γραμμή. 4207 του ιδίου υπέρ κατά εποχές απορρίπτεται. Έχουμε τώρα ένα πιλωτικό πρόγραμμα που θα το δούμε αύριο με τα υπόλοιπα. Και ερχόμαστε στην Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Υποστήριξη το Άσυλο. 4208 χάρτων ψηφί υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 449 ο εισηγητής. Η εισηγήτρια, συγγνώμη, είναι υπέρ. Α, εμένα μου είχαν πει ότι είναι κατά. Άλλος υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Το suivant est également adopté puisqu'il est identique. Και η επόμενη ταυτίζεται. Πάμε στο επόμενο. Στον τίτλο 3 συνεισφορά 4208 χάρτονγκ. Ψήφι υπέρ. Κατά. Άποχες. Νομίζω ότι είναι η ίδια πλειοψηφία υπέρ, κατά. Άρα εγκρίνονται αυτές τις τροπολογίες. Στη συνέχεια έχουμε πάλι πιλωτικά προγράμματα. Πάμε στην 4210 του κυρίου Χάρτον, ψήφι υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. Για την Ευρωπαϊκή Αστυνομική Υπηρεσία, στο τίτλο 3. 4210 Χάρτον, απορρίπτεται. 4562 Γιώτα Χάου, εισηγήτρια υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Ευρωπαϊκή Αστυνομική Ακαδημία 42-11 χάρτων υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Η επόμενη έχει αποσυρθεί. Επόμενη πίστοση πάλι χάρτων υπέρ 42-11 κατά αποχές απορρίπτεται. 899 από την Ευρώπη της Ελευθερίας και της Δημοκρατίας. Συγήτρια κατά ψήφι. υπέρ Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Και η επόμενη. 454 3 υπέρ, ψήφι υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Και η επόμενη επίσης ε, εγκρίνεται. Επόμενη σελίδα. Πρόληψη και τα λοιπά για την τρομοκρατία. 4601 Βέρτμαν, εισηγήτρια κατά ψήφι υπέρ. Κατά. Άποχες απορρίπτεται. 455 εισηγήτρια είναι κατά ψήφι υπέρ. Υπέρ. Κατά. Απορρίπτεται. Μόνο το έλκυν υπέρ αυτής της τροπολογίας. Στην 6.20. Πρώτα τα ποσά. Η συγκήτρια υπέρ. Merci, contre. Merci, abstention. Υπέρ κατά, ευχαριστώ, αποχές, εγκρίνεται. Για τα σχόλια. 620. Le rapporteur est pour. Ο εισηγητής, η συγγνώμη, είναι υπέρ, άλλη υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Και η 42-53 είναι ταυτόσιμη. Εγκρίνεται λοιπόν. Ε, το Κέντρο Παρακολούθησης Ναρκωτικών και Τοξικομανίας έχουμε την τροπολογία Βαντάλεν που δεν έχει αποσυρθεί, είναι 44-70, η συγγήτρια είναι κατά. Ψήφι κατά αποχές απορρίπτεται. Αυτή ήταν που ψηφίσαμε. Η 4470 δεν ήτανε. Όχι, η Αν. Δεν κατάλαβα ποια ψηφίσαμε τώρα. Την 462 την ψηφίσαμε. Εγώ φταίω, λέει ο πρόεδρο. Την περάσαμε, την αφήσαμε. Γιατί ε, η ομάδα μου θέλει να ζητήσει τη ψηφοφορία για τα σχόλια. Αλλά θα επανέλθουμε σε αυτό. Δεν θα πρέπει να ψηφίσουμε πρώτα τα ποσά. Ζητώ συγγνώμη, λέει ο πρόεδρο. Επανέρχομαι. Κάτι ξέχασα. Εγώ φταίω. Ξέχασα τη γραμμή πρόληψη και καταπολέμηση της εγκληματικότητας. Ε, ε, η μαφία με συμβούλευσε να το ξεχάσω αυτό, να το παρακάμψω, έτσι, ήταν εκ του πονηρού. Λοιπόν, εδώ έχουμε τροπολογίες μόνο για τα σχόλια. Όχι, είναι και για τα ποσά. Α, μάλιστα, ωραία, πολύ καλά. Δεν λέω τίποτα. 462. Πρώτα τα ποσά λοιπόν. Η συγκήτρια είναι υπέρ. Άλλη υπέρ τη καταπολέμηση εγκληματικότητα. Κατά των ποσών αυτών. Αποχές. Άρα εγκρίνεται το ποσό. 42-53 πάλι τα ποσά. Είναι το ίδιο κονδύλι και καλύπτεται από την προηγούμενη. Ωραία, καταπίπτει λοιπόν αυτή. Τώρα ας περάσουμε στα σχόλια για την 462. Η συγκήτρια είναι υπέρ. Όχι, η Γένσεν. Εκεί θέλει η ομάδα μου χωριστή ψηφοφορία, διότι θα θέλαμε να ψηφίσουμε πρώτα το τμήμα που αναφέρεται και στην αποκατάσταση ε, των ε, πρώην κρατουμένων, των ανηλίκων και τα λοιπά, ε, ΣΔΙΤ, στατιστικές, είναι ένα μεγάλο κομμάτι αυτό. Και αυτό θέλουμε πρώτο και μετά το, το επόμενο κείμενο για την πρόληψη εγκληματικών δραστηριοτήτων μετακινούμενων εγκληματικών ομάδων σε παραμεθόριες περιοχές. Θέλουμε δηλαδή χωριστά να ψηφίσουμε αυτό το θέμα της πρόληψης των ε, μετακινημένων εγκληματικών ομάδων με δραστηριότητες στις παραμεθόριες περιοχές. Αυτό το κομμάτι να ψηφιστεί χωριστά. Bon. Que tout le monde a... Μάλιστα. Καταλάβατε όλοι τη διάκριση ανάμεσα στα δύο τμήματα, αυτό που λέει Άννα Το καταλάβατε όλοι. Μάλιστα. Για το πρώτο τμήμα λοιπόν. Εισηγήτρια είναι υπέ, Για το πρώτο σχόλιο. Αυτό που δεν αρέσει στην Αν. Ψήφι υπέ, Κατά. Η φιλελεύθερη λοιπόν και η κυρία Ανδρέασεν. Αποχές. Μία. Εγκρίνεται το πρώτο τμήμα. Το δεύτερο τμήμα τώρα. Η συγγήτρια είναι υπέρ, άλλη υπέρ. Αποχές μεγαλύτερη πλειοψηφία. Εγκρίνονται και τα δύο τμήματα λοιπόν. Α, με, όχι με την ίδια, με διαφορετική πλειοψηφία. Και νομίζω ότι πρέπει να ψηφίσουμε και τα σχόλια της 4253 τώρα. Όχι, καλύπτεται. Μου λέγουν ότι καλύπτεται, διότι αντιστοιχεί στο δεύτερο τμήμα της 462 που μόλις υπερψηφίσαμε. Καλώς. Άρα δεν ψηφίζουμε. Θεωρούμε ότι είμαστε εντάξει. Και προχωρούμε. Κάλυψαμε αυτό που δυστυχώς είχα ξεχάσει. Νομίζω τώρα ότι δεν ψηφίσαμε τη 4470 του κυρίου Βαντάλεν. Απορρίψαμε την προηγούμενη, αλλά δεν ψηφίσαμε την ε, 4470. Ψήφι υπέρ, η κατά. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. Οπότε περνούμε στο κονδύλι Prince. Ε, είναι η άδουσα γραμμή. Ψήφι υπέρ της 1006. Κατά. Η κατά. Αποχές ε, απορρίπτεται. 431 υπέρ. Κατά Αποχές εγκρίνεται. 4.32. Εδώ έχουμε πρώτα τα ποσά. Εισηγήτρια υπέρ. Ψήφι υπέρ. Κατά. Χρειάζεται εδώ αναγκαστικά ηλεκτρονική ε, ψηφοφορία. Αρχίζει τώρα, σας παρακαλώ. Ψηφίζουμε τα ποσά της 432. Πέρας, αξιολόγηση και εκτίμηση αντικτύπου. Με ταχύτητα φωτός ψηφίσαμε. 19 υπέρ, 20 κατά απορρίπτεται. Τα σχόλια. Έχει νόημα να τα ψηφίσουμε εφόσον ψηφίσαμε τα ποσά. Ναι. Η συγκίτρια είναι υπέρ. Άλλη υπέρ. Κατά. Νομίζω με την ίδια πλειοψηφία. Οπότε ξανά ηλεκτρονική για τα σχόλια παρακαλώ. Αρχίζει τώρα η ηλεκτρονική ψηφοφορία για τα σχόλια. Ψηφίστε σας παρακαλώ αγαπητοί συνάδελφοι, πέρας. 14 υπέρ 21 κατά απορρίπτονται τα πάντα για αυτή την τροπολογία. 4.34. Συγγήτρια είναι υπέρ. Ψήφι υπέρ. Ευχαριστώ. Κατά. Ευχαριστώ. ποχε. Α, έλεγχο. Να το επαληθεύσουμε γιατί το ΕΛΚ δεν είναι τελείω απομονωμένο στην καταψήφιση. Ευχαριστώ. Πέρας. 18 υπέρ, 20 κατά. Άρα η τροπολογία απορρίπτεται. Ερχόμαστε στη 44 ισότητα υπέρ, εισηγήτρια είναι υπέρ, κατά, αποχές 44,71, 44-71 Βαντάλεν διατηρείται, εισηγήτρια κατά, ψήφι υπέρ, κατά, αποχές απορρίπτεται. 4.35 εισηγήτρια κατά, ψήφι υπέρ, κατά, αποχές απορρίπτεται. Γυρνάμε σελίδα. 4472 Βαντάλεν εισηγήτρια κατά. Ψήφι Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 436 εισηγήτρια κατά. Ψήφι Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Η 437. Εδώ τι έχουμε. Πρώτα τα ποσά. Η εισηγήτρια είναι υπέ. Ψήφι Κατά. Αποχές. Εγκρίνονται τα ποσά. Τα σχόλια τώρα. Η συγκεκριμένη είναι υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται επίσης. Καταπολέμηση της βίας. Το πρόγραμμα Δάφνη. 10-23. Η συγκεκριμένη είναι κατά. Ψήφι υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 39. Ψήφι υπέρ. Η συγκεκριμένη υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Οι υπόλοιπε τροπολογίες θα ψηφιστούν μόνο για τα σχόλια τους. 6-19, εισηγήτρια υπέρ, ψήφι υπέρ. Κατά, αποχές, εγκρίνεται. 47-66, εισηγήτρια κατά, ψήφι υπέρ. Κατά. Αποχές. Έχουμε μια ελαφρά πλειοψηφία κατά. 43-80. Α, ταυτόσημη και άρα απερίφθη. 47-67. Εισηγήτρια κατά. Ψήφι Κατά, μάλλον χρειάζεται ηλεκτρονική επαλήθευση, θα είναι πάρα πολύ μικρή διαφορά. Ψηφίζουμε 47-67. Votons. Nous votons. Nous continuons Ψηφίζουμε, ψηφίζουμε. Άλλοι δύο που δεν ψήφισαν. Πέρας. 19 pour 16 υπέρ 16 κατά εγκρίνεται η τροπολογία. Έχουμε ένα πιλωτικό πρόγραμμα τώρα και πάμε στη Eurojust πιο κάτω και ψηφίζουμε την 438 την οποία υποστηρίζει και η συγκήτρια πρέπει να σας ψήφι υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Όπως και η επόμενη. La contribution au titre 3 d'Eurojust. Eurojust, συνεισφορά στο τίτλο 3. Ψηφίζουμε. 439 υπέρ και η συγκήτρια υπέρ είναι. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Οπότε η επόμενη εγκρίνεται και αυτή. 463. Ποινική δικαιοσύνη. Πρώτο το ποσά. Η συγκήτρια είναι υπέρ. Υπέρ των ποσών κατά. Αποχές εγκρίνεται. Τα σχόλια. Η συγκήτρια είναι υπέρ. Άλλη υπέρ κατά, φιλελεύθερη, κύριος Χάρτον κλπ. Αποχές εγκρίνεται επίσης. Τώρα έχουμε πιλωτικό πρόγραμμα, γυρίζουμε σελίδα και φτάνουμε σε άλλο πρινς. Χώρος ελευθερίας, ασφάλεια και δικαιοσύνης. 10.24 της Γκουα εισηγήτρια κατά, ψήφι Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 4.40 η συγγήτρια είναι υπέρ, υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Στην 441, πρώτο το ποσό. Η συγγήτρια είναι υπέρ, άλλη υπέρ, κατά, α, α, α, ηλεκτρονικά για την 441 το ποσό. 4-41. Άρχεται η ψηφοφορία. Παρακαλώ ψηφίστε συνάδελφοι. Πέρας. Ψήφισαν όλοι. 18 υπέρ, 20 κατά. Απορρίπτονται τα ποσά. Απορρίπτονται τα ποσά. Τα σχόλια ισχύουν. Να ψηφίσουμε τα σχόλια τουλάχιστον. Υπέρ των σχολείων. Ναι, Κατά. Η ίδια πλειοψηφία. Απορρίπτεται επίση η τροπολογία 441. Έχει εξολοθρευτεί πλήρω. Αλλά μπορεί να ξανάρθει στην Ολομέλεια. Αν το επιθυμείτε. Τελειώσαμε λοιπόν με το 3-1. Πάμε στο 3Β. Όχι, δεν είστε έτοιμοι. Στο 4. Ούτε γι' αυτό είστε έτοιμοι. Πέντε. 5 3. τμήμα τρίτων, Ο προπολογισμό τη Κομισιόν. πέντε Μπαλζάνη. Πάρτε το έγγραφο πέντε. Α, κάνουμε μικρή διακοπή δύο λεπτών. Είμαστε σε πλήρη φόρμα και σε ρυθμό έχουμε παλμό και μπορούμε να συνεχίσουμε και να τελειώσουμε απόψε, δεν υπάρχει λόγος να στερήσουμε από τον εαυτό μας αυτή τη χαρά. Bon. Je minutes pour que... Διακόπτω δύο λεπτά για να κοιτάξουν οι ε, συνεργάτες αν μπορούμε να ψηφίσουμε το έγγραφο 5, τον τίτλο 5, μόνο για την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Διακοπή 10 λεπτών. Διότι οι πολιτικές ομάδες πρέπει να κάνουν φωτοτυπίες στις λίστες ψηφοφορίας για τον τίτλο 5. Θυμίζω ότι ε, ψηφίζουμε μόνο την ε, κατηγορία 5 της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, γιατί για τα υπόλοιπα θεσμικά όργανα δεν έχουν ολοκληρωθεί οι πολιτικές συμφωνίες. Voilà, mes chers collègues, est-ce qu'on peut reprendre... Λοιπόν, αγαπητοί μου συνάδελφοι, μπορούμε να συνεχίσουμε. Voilà, je vous demande de reprendre déjà vos places. Σας παρακαλώ καθίστε. Un, Encore un peu de temps. Η συγκήτριά μας έχει ε, λίγο περισσότερο χρόνο να ζητήσει.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 Voilà, il faut peut-être euh, oui, récupérer ceux de nos collègues. Λοιπόν, θα πρέπει να ξαναφωνάξουμε τους συναδέλφους μας που βρήκαν την ευκαιρία να πάνε να πιούν ένα περιτύφ ή ένα τσάι, εν πάση περιπτώσει. Διότι δεν θα πρέπει τώρα να έχουμε προβλήματα στις ψηφοφορίες. Τώρα που ετοιμάζεται η συγγήτρια, σας θυμίζω ότι θα ψηφίσουμε το τίτλο 5 μόνο για το προϋπολογισμό της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, κατηγορία 5. Έτσι δεν είναι? J'en profite pour poser Α, σας ρωτάω και για την κατηγορία 3β επευκαιρία και μου λέγουν ότι το Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα δεν είναι έτοιμο να ψηφίσει για την 3Β και προτιμάει να περιμένει μέχρι αύριο, έτσι είναι. Bon. Je τι είναι αυτά τα χαμόγελα από το ΕΛΚ, ε, προς επίρρωση είναι τον όσο λέω, μάλιστα. Ήρισε και η Μπάρμπαρα, άρα μπορούμε να ψηφίσουμε. est d'accord pour voter. Πάντως για τον τίτλο 5 για την Ευρωπαϊκή Επιτροπή συμφωνείτε όλοι να ψηφίσουμε, έτσι. Donc, euh, téléphoner, euh. Είναι ακόμα άδεια κάποια έδρα, δεν τους παίρνετε τηλέφωνο. Madame le rapporteur. Η συγγήτρια. Είσαι έτοιμη, Φραντσέσκα. Prête, on peut commencer On peut commencer. Donc... Μπορούμε να αρχίσουμε να ψηφίσουμε. Τον τίτλο 5 ψηφίζουμε, λέει η συγκήτρια. So, sorry. Please. Eh, adesso quindi possiamo procedere al voto della rubrica 5. Πρέπει να προχωρήσουμε στην ψηφοφορία του τίτλου 5. 3β αύριο το πρωί. Εντάξει, ωραία. Μάλιστα, ολοκληρώνουμε απόψε με την κατηγορία 5, τίτλο 5. Euh, Εάν συμφωνεί η συγγετρία, σας προτείνω να δείτε τον πίνακα που υπάρχει στο συμπληρωματικό φάκελο για τις ψηφοφορίες ή στον προϋπολογισμό Στη σελίδα Τροπολογίες της επί τίτλος 5. Έχει μόνο μια σελίδα και λέει ότι εδώ είναι όλες οι γραμμές και ότι μπορούμε και ενδεχομένως να ψηφίσουμε μπλοκ. Πρόκειται για την αποκατάσταση του προπολογισμού, του σχεδίου που μάλλον προπολογισμού της Κομισιόν. Alors, Όλοι έχετε αυτόν εδώ το πίνακα που δείχνει ο Πρόεδρος. Εμεί, όχι πάντως. Έχετε αυτό εδώ το έγγραφο. Πρέπει όλοι να το έχετε πριν να ψηφίσουμε. Ça, ça marche Δυστυχώς οι σελίδες δεν είναι αριθμημένες, λέει ο Πρόεδρος. Ο... Λέει, τροπολογίες της εισηγήτριας, τίτλος 5, Κομισιόν. Η Γενική Εισηγήτρια λέει ότι όλες μαζί είναι στον τίτλο 5, κατηγορία 3. Προτείνω να ψηφίσουμε unblock, εκτός αν κάποιος ζητήσει χωριστή ψηφοφορία κατά τμήματα, η εισηγήτρια. Ήθελα μόνο να διευκρινίσω ότι αυτή η αποκατάσταση του σχεδίου προπολογισμού της Κομισιόν δεν λαμβάνει υπόψη το 2, την ε, διορθωτικό προπολογισμό 2 που σχετίζεται με την Κροατία. Και είναι εκτός αυτό της αποκατάστασης δηλαδή. D'accord. Sur lequel y aura un autre vote. Γι' αυτό θα κάνουμε χωριστή ψηφοφορία. Μάλιστα. Για επ' αυτού θα μιλήσουμε με το Συμβούλιο κατά τη συνδιαλλαγή. Είναι μια διορθωτική επιστολή που δεν ψηφίστηκε από το Συμβούλιο και θα το συζητήσουμε με το Συμβούλιο τη στιγμή της συνδιαλλαγής. Ωραία. Λοιπόν, αποκατάσταση του σχεδίου προϋπολογισμού χωρίς να λάβουμε υπόψη τις αλλαγές που προτείνει το διορθωτική επιστολή. Όλοι είστε σε θέση να ψηφίσετε. Ψηφίζουμε λοιπόν unblock. Ποιοι είναι υπέρ. Ευχαριστώ. Κατά. Δύο. Αποχές. Δεν υπάρχουν αποχές και εκτιμούμε το χαμόγελο στα πρόσωπα των εκπροσώπων της Επιτροπής. Αλλά τώρα θα ψηφίσουμε τα αποθεματικά, γιατί όλα αυτά θα τα βάλουμε σε αποθεματικό. Τέρμα τα χαμόγελα. τώρα... <laughs> Θα ξαναπάρουμε το εγγραφάκι μας και κατηγορία 5 αρχίζει στην σελίδα 198 και τα αποθεματικά τα έχουμε. Καταρχήν έχουμε μια γραμμή που δεν καλύπτεται από αυτή την ψηφοφορία unblock που είναι στη σελίδα 202. Είναι τοπικό προσωπικό της Διεύθυνσης ε, Επικοινωνίας. Η 4426 του κυρίου Φαντάλεν. Ε, η συγκίτρια είναι κατά. Ποιοι είναι υπέρ. Κανείς. Ένα, δύο, δύο, τρει-τέσσερι Κατά. Ευχαριστώ. Αποχές. Απορρίπτεται. Στη συνέχεια Γυρνάμε τις σελίδες και περνάμε στις θέσεις αποθυματικό για την 496. Ε, η συγκήτρια είναι υπέρ. Ποιοι είναι υπέρ. Κατά. πρέπει να επαληθεύσουμε. Νομίζω πως υπάρχει μια πλειοψηφία κατά, αλλά επαληθεύουμε ηλεκτρονικά. Αρχίζει η ψηφοφορία για τη θέση αποθεματικό της, 400, της 496. Ψηφίστε αγαπητοί συνάδελφοι. Ah, je vois qu'il y a des renforts qui arrivent. Les renforts pour les mises en réserve. Voilà, Le vote est... Le vote est... Oui, oui, le vote est clos. Τέλος της ψηφοφορίας. 20 κατά, 17 υπέρ απορρίπτεται. Οπότε η Κομισιόν το χαμόγελο της έχει φτάσει στα αυτιά. 621. Η συγκίτρια είναι υπέρ. Ποιοι είναι ε, υπέρ, κατά. Νομίζω έχουμε την ίδια πλειοψηφία, αλλά θα επαληθεύσουμε για την 621. Ψηφίστε αγαπητοί συνάδελφοι, δεν ψηφίσατε όλοι. Ψηφίσατε τώρα όλοι. 16 υπέρ, 21 κατά. Η ίδια διαφορά. Οπότε απορρίπτεται. 43-78 απορρίπτεται και αυτό. Περνάμε τώρα στην επόμενη γραμμή. Α, κύριε Άρτογκ. page. Yes. Alors, euh, la page est la page 205. En haut de la page 205. L'amendement 514. Πάνω πάνω στο 205. Τροπολογία 214. Όχι, 540. Λάθος, συγγνώμη. Θέση σε αποθεματικό. Η συγκίτρια είναι υπέρ, ποιοι είναι υπέρ, κατά. Η ίδια πλειοψηφία αποχές απορρίπτεται. Τροπολογία 43.00. Η εισηγήτρια είναι κατά. Ποιοι είναι υπέρ. Κατά. Πολύ διασκεδαστικό. Αντίστροφη πλειοψηφία φαίνεται και προτιμώ να επαληθεύσουμε. Είναι για την IT. Άρχεται η ψηφοφορία. Αγαπητοί συνάδελφοι, ψηφίστε. «18 υπέρ, 17 κατά, εγκρίνεται». 515. Ποιοι είναι υπέρ, η συγκίτρια είναι υπέρ. Ποιοι είναι υπέρ. Κατά. ηλεκτρονική ψηφοφορία λυπάμαι, αλλά είναι παράξενο ότι παθιάζουν πολύ περισσότερο τα αποθέματα από ότι τα νούμερα. Τέλος της ψηφοφορίας. 16 υπέρ 19 κατά απορρίπτεται. Γυρνώ σελίδα τώρα και φτάνω στην 207, στα μέσα της 207 Ψηφιακές δημοσιεύσεις. 348. Η συγκίτρια είναι κατά. Ποιοι είναι υπέρ. Κατά. Λυπάμαι για το ΕΛΚΑ. Αυτή η 348 απορρίφθηκε. Κάτω-κάτω στη σελίδα έχουμε μια τροπολογία 42 85 Σαλβατόρ Γκαρίγκα την έχει υπογράψει. Τη αποσία του θα τον τιμήσουμε υποστηρίζοντα αυτή την τροπολογία. Η συγγήτρια είναι υπέρ. ποιοι είναι υπέρ. Κατά. Αποχές. Να συγχαρούμε τον Σαλβαντόρ για αυτήν την ομόφωνη υπερψήφιση της τροπολογίας του. Είναι θέση σε αποθυματικό. Γυρνάμε σελίδα. J'en 210, 211 et le... Σελίδες 210 και 211 και πάνω πάνω στην 212. Μέχρι τον τίτλο που λέει βιώσιμη ανάπτυξη. Χωρίς τη βιώσιμη ανάπτυξη. Έχουμε εδώ μια σειρά τροπολογιών, σε δυόμιση σελίδες είναι αυτές που πρέπει να τις ψηφίσουμε Ο Πρόεδρος, σας προτείνω το εξής. Έχουμε πάνω πάνω στη σελίδα 2.10 δύο τροπολογίες που ξεπερνούν το σχέδιο προπολογισμού. Οπότε θα τις ψηφίσουμε ξεχωριστά. Στη συνέχεια θα υποβάλω μπλόκ τις άλλες τροπολογίες που αποκαθιστούν το σχέδιο προπολογισμού. Είναι λογικό. 465 που είναι πάνω από το σχέδιο προϋπολογισμού. Ποιοι είναι υπέρ. Σας ευχαριστώ. Αποχές εγκρίνεται. 4571 Utah Haug. Ποιοι είναι υπέρ. Κατά. Αποχές είναι το ίδιο. Αυτά τα δύο εγκρίνονται λοιπόν. Τώρα ψηφίζουμε μπλοκ όλη την υπόλοιπη σελίδα 2.43 στα ελληνικά 2.44 και την 2.45 μέχρι ε, τελευταία τροπολογία της Χαόγκ είναι η 45.74 Ποιοι είναι υπέρ, κατά αποχές εγκρίνονται στη συνέχεια Μπορούμε να γυρίσουμε σελίδα. Πάμε δηλαδή στη 246 στο ελληνικό κείμενο. Είμαστε στην γραμμή ε, δαπάνες των θεσμικών οργάνων και έχουμε την 4301 για θέση αποθεματικό και η συγκίτρια είναι κατά. Δαπάνες διαχείρισης οργάνου. Ε, θα ψηφίσουμε ηλεκτρονικά για επαλήθευση. 4301 είναι κάτω-κάτω σελίδα 247 στο ελληνικό κείμενο. Αρχίζει η ψηφοφορία, τέλος της ψηφοφορίας. 20 υπέρ, 16 κατά, εγκρίνεται. Αυτή η γραμμή λοιπόν μπαίνει σε αποθηματικό. 534. Η συγγήτρια είναι υπέρ. Ποιοι είναι υπέρ. Κατά. Να επαληθεύσουμε ηλεκτρονικά. Κλείστε την ψηφοφορία και ξανανοίξτε την ψηφοφορία. Λοιπόν, 534 ψηφίζουμε τώρα. Η συγκίτρια είναι υπέρ. Ψηφίσατε όλοι. Τέλος ψηφοφορίας. Μπράβο, είστε γρήγοροι. 17 υπέρ, 19 κατά. Αυτή τη φορά απορρίπτεται. Στη συνέχεια περνάμε στη γραμμή συνεδριάσεις των Επιτροπών. Η εισηγήτρια είναι υπέρ. Υπέρ, κατά. Ίδια πλειοψηφία, αλλά σε επαληθεύσουμε. Την 534 ψηφίζουμε λοιπόν ηλεκτρονικά. Le vote est ouvert, le vote Τέλος της ψηφοφορίας απορρίπτεται. 43.01. Η συγκίτρια είναι κατά. Ποιοι είναι υπέρ? Vote électronique. Ηλεκτρονική ψηφοφορία. Νομίζω πως η πλειοψηφία είναι υπέρ, αλλά ψηφίζουμε ηλεκτρονικά. Ψηφίσατε όλοι, 21 υπέρ, 16 κατά. Εγκρίνεται λοιπόν αυτό το αποθυματικό. Très bien. Euh, euh, Τελειώσαμε. Τα αποθεματικά για το προσωπικό είναι σε μια γραμμή χ, χ, χ. Δεν ξέρω τι θα πει αυτό, αλλά εσείς καταλάβατε. Και εδώ θα σταματήσουμε γιατί τα άλλα τμήματα είναι ήδη το κοινοβούλιο. Αγαπητοί μου συνάδελφοι, λοιπόν, ε, τελειώσαμε νωρίτερα. Είστε βέβαιοι ότι το 3β δεν είναι δυνατό να το τελειώνουμε. Ο Γκαρίγκα δεν είναι εδώ. Μάλιστα. Λοιπόν, σας ευχαριστώ. Σας συγχαίρω. Νομίζω ότι η καλή συνεννόηση ανάμεσα στις ομάδες και η συνεργασία ανάμεσα στους διάφορους ε, αρμόδιους επιτρέπει να προχωρήσουμε πολύ γρήγορα και δεν αποκλείω ότι μπορεί να τελειώσουμε τις ψηφοφορίες αύριο στο τέλος του πρωινού. Πριν να τα χωρίσουμε όμως, μήπως μπορούμε να ψηφίσουμε την έκθεση Καλφίν τώρα. Κρίμα, κρίμα. Μία μόνο ψήφο, ψηφοφορία και θα είχαμε ξεμπερδέψει. Μπάση περιπτώσει, αύριο το πρωί θα ξαναρχίσουμε με τη σειρά που προβλεπόταν και θα έχουμε στόχο να τελειώσουμε όσο γίνεται πιο γρήγορα. Θα έχουμε στόχο να τελειώσουμε αύριο το απόγευμα και δεν αποκλείται να τελειώσουμε και αύριο το μεσημέρι. Πάρα πολύ ωραία. Πέρα συνεδρίασης.